από τις ομάδες των σοσιαλιστών και των, του ECR και του μία εγγεγραμμένων ε, έλαβα κάποια αιτήματα τροποποίησης ε, των μελών που συμμετέχουν στις ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Θα ε, συμπεριληφθούν αυτά στα πρακτικά και αν δεν υπάρξει κάποια παρατήρηση ή ένσταση μέχρι την έγκριση των πρακτικών θα εγκριθούν αυτές οι τροποποίησεις.